συνεργασίας στο πλαίσιο της ε, Στοκχόλμης πάντοτε. Ε, λίγη συζήτηση, ευχαριστούμε Επίτροπε. Η ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον συντάκτη της προφορικής ερώτησης, τον συνάδελφο Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, τα ερωτήματα που σας θέτω εξ ονόματος της Επιτροπής αφορούν το μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τη δυνατότητα δηλαδή να επέμβουμε σε αυτή τη δομή για να διορθώσουμε τα ελλείμματα και τα προβλήματα που έχει και με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στην εσωτερική αγορά. Όπως ξέρετε και εσείς και οι συνάδελφοι, η Συμφωνία για τη Δημιουργία του ΕΟΧ ανάγεται στο 1994, άρα ε, υπάρχουμε, έχει, έχουμε πίσω μας ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να κάνουμε μια αξιολόγηση. Ε, ε, είναι μια συμφωνία που συνήθει ανάμεσα στις χώρες ΕΖΕΣ και την ε, ευρωπαϊκή κοινότητα, ούτω ώστε οι χώρες ΕΖΕΣ να μπορούν να συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά και στις σχετικέ δραστηριότητε χωρίς να γίνουν μέλη της ΕΟΚ. Τώρα έχουμε μια καινοτομία απέναντι μας που δεν σχετίζεται μόνο με τον πιθανό έλεγχο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΕΟΧ, αλλά έχει να κάνει με το αίτημα ορισμένων μικρών ευρωπαϊκών χωρών και πιο συγκεκριμένα την Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό, που θέλουν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μικρές χώρες, αλλά ε, που έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και που θέλουν σαν προοπτική να ε, ενταχθούν στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή στις δομές της και στην θεσμική της διάσταση. Τι πρέπει να κάνουμε. Η Κομισιόν ανέφερε δύο δυνατότητες. Η πρώτη, όπως ξέρετε, είναι να δημιουργηθεί μια συμφωνία πλαίσιο σύνδεσης μεταξύ αυτών των χωρών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η δεύτερη λύση είναι η προσχώρηση αυτών των τριών μικρών κρατών απευθείας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα που ονομάζεται Ελβετία. Η Ελβετία είναι η μοναδική χώρα που αυτή τη στιγμή είναι κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, που ποτέ επίσημα δεν μπήκε στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο λόγος, όπως θα θυμάστε πολύ καλά, είναι το αρνητικό αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος μεταξύ των Ελβετών πολιτών. Εμείς έχουμε ένα αντικειμενικό συμφέρον να δικτυώσουμε όλες αυτές τις δομές μεταξύ τους και να δώσουμε μια δυνατότητα ε, θετικής και αποτελεσματικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις πιο μικρές από αυτές τις χώρες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε, ποιο δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, ούτω ώστε να μην την αχθεί στον αέρα λόγω της Ελβετίας η πολύ επικοδομητική σχέση που αποδείχθηκε ότι έχουμε με τη χώρα αυτή ε, μέσω διμερών συμφωνιών. Πάνω από 120 τέτοιε διμερεί τομεακέ συμφωνίε υπάρχουν ανάμεσα στην Ελβετία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτουμε λοιπόν ερωτήματα που είναι ρητορικά στην πραγματικότητα, γιατί προποθέτουν ποια είναι η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί σε αυτέ τι ερωτήσει. Ρωτάμε λοιπόν, δεν κρίνει η Επιτροπή ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή, όπω έλεγα προηγουμένω, να εξεταστεί η λειτουργία τη συμφωνία του ΕΟΧ που ισχύει από το 1994, γιατί πέρασαν ήδη από τότε σχεδόν 30 χρόνια. Ε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να πούμε αν ε, το πείραμα αυτό υπήρξε θετικό ε, ή αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, κάποια προβλήματα. Αυτά τα χρόνια ήταν γεμάτα γεγονότα. Και από τα γεγονότα αυτά μπορούμε να αντλήσουμε τις ενδείξεις ούτω ώστε ενδεχομένω να διορθώσουμε τη συμφωνία ίδρυση του ΕΟΧ και να την ενισχύσουμε. Σας ρωτάμε λοιπόν, έστω και έμεσα, ανάμεσα στις δύο αυτές εναλλακτικέ επιλογές που μας ε, παρουσιάσετε, κατά τη γνώμη σα ποια θα ήταν πιο αποτελεσματική. Ούτως ώστε να αξιοποιηθεί περισσότερο ο ΕΟΚ σχεδόν 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Το δεύτερο ερώτημα που συνδέεται στενά με το προηγούμενο είναι το εξή. Θεωρείτε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον αντίκτυπο πάνω στην ενιαία αγορά που θα είχε η ενδεχόμενη διεύρυνση της συμφωνίας του ΕΟΚ ούτω ώστε να συμπεριλάβει και αυτέ τι χώρε που ανέφερα προηγουμένω. Θα μπορούσαν να μπουν επίσημα οι τρει αυτέ χώρε στον ΕΟΧ και να έχουν στενή σχέση μέσω αυτού του εργαλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΖΕΣ χρονολογείται από το 1960. Είναι πάρα πολύ παλιά, αρχαία ε, αυτή η συμφωνία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω α, αυτή την έκφραση. Ε, Όμω δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τη συμφωνία αυτή γιατί έχουμε αυτή την ιδιαίτερη σχέση με την Ελβετία. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα στον ΕΟΧ, που είναι μια συμφωνία πιο πρόσφατη, που είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και να επικαιροποιηθεί ε, υπό το φως της εμπειρίας που έχουμε συγκεντρώσει και έτσι ο ΕΟΧ θα μπορούσε πολύ άνετα να συμπεριλάβει την Ανδόρα, το Άγιο Μαρίνο και το Μονακό περιμένοντας ε, περαιτέρω πλησίασμά τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας έλεγα λοιπόν, με τις ερωτήσεις που κάνουμε δείχνουμε έμεσα ποιες είναι οι προτιμήσεις μας, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κοφεράτη, Επίτροπος κυρία Μάλιστο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας με τη σειρά τους. Όπως γνωρίζετε, η Συμφωνία Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έτυχε διαπραγματεύσει πριν από 20 χρόνια και οι συνθήκε ήταν διαφορετικέ από τις σημερινέ. Τα συμβαλόμενα μέρη γνωρίζουν το ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον. Συνεπώ, πολύ καλή είναι η αναθεώρηση τη λειτουργία τη συμφωνία ε, που δημοσιεύτηκε από την Νορβηγία, τον Χθεστάν και την Κομισιόν πέρσι τον Δεκέμβρη. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία εξακολουθεί να λειτουργεί ε, σε εγκαίες ικανοποιητικά. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες ε, των τριών χωρών ε, ΕΖΕΣ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να μειώσουν τον αριθμό των νομικών πράξεων πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία ε, αλλά είναι σημαντικό οι χώρε τη να το θέσουν ω προτεραιότητα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι αρχέ τη ομογένεια και τη νομική ασφάλεια ε, εγγυώνται την αποτελεσματικότητα, την βιωσιμότητα και την αξιοπιστία τη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν γνώμονα όλων των συμβαλωμένων μερών η αύξηση της χορήγησης αρμοδιοτήτων σε ε, υπηρεσίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής θα πρέπει ε, να απηχηθεί και στον ε, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι οικονομικές πράξεις που δημιουργούν αυτά τα όργανα προβλέπουν τη συμμετοχή και τρίτων χωρών, σήμερα βλέπουμε το χωρών ΕΖΕΣ και του ενίου οικονομικού χώρου, ως παρατηρητών. Προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Ε, για παράδειγμα, η περιοχή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τι χώρε ΕΖΕΣ εξαιτία των εξουσιών που δίδονται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ε, η αρχή επιτήρηση ε, τη ΕΖΕΣ. στη δομή των δύο πυλώνων η, αυτή η επιτροπή παίζει το ρόλο της Κομισιόν. Όμως, όταν έχουμε θέματα προστασία τίμων σε οικονομικούς φορείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφορετική προσέγγιση από την ε, ΕΖΕΣ ε, για το κατά πόσον ε, η Επιτροπή της ΕΖΕΣ θα πρέπει να έχει τις ίδιες εξουσίες που έχει η Κομισιόν. Να μπορεί να επιβάλλει δηλαδή πρόστιμα σε οικονομικούς φορείς. Επίσης, ρωτήσατε για την Ανδόρα, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο και τη διεύρυνση. Η Κομισιόν πέρσι υιοθέτησε μια ανακοίνωση σε σχέση με αυτούς τους τρεις ε, γείτονε με πέντε εναλλακτικά σενάρια για τη συμμετοχή τους α, ξεκινώντας από το πιο φιλόδοξο στο λιγότερο φιλόδοξο. Το, πέρσι το Δεκέμβρη το Συμβούλιο ζήτησε περαιτέρω ανάλυση από τη βάση δύο από, από αυτά τα σενάρια. Ε, πρώτον, η συμμετοχή αυτών των τριών χωρών στο ε, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ε, δεύτερον ε, ε, συμφωνίες ε, συνεργασίας με αυτές τις ε, χώρες, μία ή περισσότερες συμφωνίες για την συμμετοχή τους με θεσμικούς μηχανισμούς σύμφωνα με, με τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου. Ε, επεξεργαζόμαστε αυτή την έκθεση την οποία θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πριν το τέλος του χρόνου με συστάσεις για τα επόμενα βήματα οι πιθανές επιπτώσεις της συμμετοχής αυτών των τριών χωρών στην, Ευρω... στο... στην αγορά αναλύεται αυτή τη στιγμή, αλλά εξαιτία του μικρού πληθυσμού τους μάλλον θα είναι πολύ μικρές αυτές οι επιπτώσεις. Μιλάμε για περίπου 150.000 άτομα μόνο. Παρ' όλα αυτά, είναι κανόνες και η σωστή εφαρμογή τους είναι σημαντική ε, για να... Ε, για την ε, εξασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός. Τώρα, Ελβετία. Ε, δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκό ομονίες Χώρος λειτουργεί καλά, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή της Ελβετίας αυτών θα ήταν η πιο απλή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Η διεύρυνση της έννοιας αγοράς ε, στην Ελβετία θα ωφελούσε τους καταναλωτές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελβετία θα, είναι, θα διευκολυνθεί ε, η κυκλοφορία των προϊόντων και θα βελτιωθεί, θα, αυξηθεί, ε, θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής ε, των πολιτών μας. Ε, η σημερινή προσέγγιση, η τομιακή προσέγγιση, δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμή των κανόνων της ενίας αγοράς. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αν η Ελβετία αποφασίσει να ε, προσχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα βρούμε μια άλλη λύση θεσμική. Ετοιμαζόμαστε για ε, διαπραγματεύσει με την Ελβετία σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε μέγιστη διαφάνεια και νομική ασφαλεία για τους καταναλωτές και τους, ε, και τις επιχειρήσεις στην ε, εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο Ανδρέας Σφάπ, εκ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, προχωρημένη ώρα. Πάντως χαίρομαι που έρχεστε για να απαντήσετε με τόσο αφή τρόπο τα ερωτήματα της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Ο Σάνφος Σάντσες Σμιτ θα εμβαθύνει. Εγώ θα επικεντρωθώ τώρα στην Ελβετία που αναφέρατε και στο τέλος τη κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Κοφεράτη στην εισαγωγική του παρέμβαση είπε ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής με την ε, Ελβετία έχει ο ίδιος ενδιαφέρον να ενημερώνετε βέβαια για το πώς βαίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εσείς είπατε ότι στο θεσμικό πλαίσιο μιας ε, συμφωνίας θα Προσπαθήστε να αναπτύξετε μια συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έστω και χωρί την Ελβετία. Μια διμερή συμφωνία, ωστόσο, στο πλαίσιο του, του δικαίου του ανταγωνισμού, δεν θα ήταν μια σκόπιμη προσπάθεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προσφερθεί μια θεσμική λύση στην Ελβετία. Μια ρεαλιστική λύση. Και φαντάζομαι ότι και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα έχει ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό και θα αναπτύξει κάποιο σενάριο αλλά έστω από εσά για την ενέργεια τουλάχιστον μπορείτε να μα πείτε τι έχει μέχρι τώρα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια περαιτέρω εδραίωση μια συμφωνία ε, με την Ελβετία για την ενέργεια και σε ποιο βαθμό μπορεί να το δέχεται αυτό η Ελβετία. Για τα δε τα διαφιλονικούμενα ζητήματα τα οποία υπάρχουν έστω και ολίγα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετίας. Υπάρχουν ρυθμίσει, ή λύσει μέσα σε ένα νομικό πλέγμα που να είναι αποδεκτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ελβετία με την αποδοχή ενός εντό εισαγωγικών ε, ξένου δικαστή, αλλοδαπού δικαστή. Ευχαριστώ. Άδελφος Ερτούκ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, τόσο ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος όσο και οι διμερείς 120 αριθμό συμφωνίες που έχουμε με την Ελβετία δείχνουν πόσο ελκυστική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και για κράτη εκτός αυτής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως κράτη ε, είναι υποχρεωμένα βεβαίως να ε, ικανοποιούν ευαισθησίες των πολιτών τους όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία παραδείγματι που ξέρουμε ότι έχει προσπαθήσει η Ισλανδία δύο φορές η Νορβηγία δύο φορές ε, και δεν μπόρεσε λόγω δημοψηφίσματος το οποίο απάντησαν αρνητικά οι πολίτες και η Ισλανδία λόγω των οικονομικών δυσχεριών που πέρασε αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το όνειρο της ένταξης Ευρωπαϊκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη ε, ίσως ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ε, να αποτελεί μια ικανοποιητική λύση και κυρίως για τα τρία μικροκράτη, τα πολύ μικρά κράτη, τα οποία ίσως να βρουν εκεί κατάλληλο πεδίο δράσης. Ε, ρωτώ λοιπόν την Επίτροπο κυρία Μάλστρομ. Υπάρχει δυνατότητα να έχετε τη δυνατότητα να μας μιλήσετε, για τα τρία αυτά πολύ μικρά κράτη να, να ρυθμιστούν οι σχέσεις μας μαζί τους. Συνάδελφος Βίλαν. Ευχαριστώ. Στον ΕΟΧ υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, κεφαλαίου, ε, προσώπων ε, και αυτό το σημαίνει ότι μεταφέρεται το κοινοτικό κεκτημένο και στις ε, τρίτες χώρες. Ε, έχουν υποχρέωση, παραδείγματος χάρη, για την ε, προστασία του καταναλωτή. Το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως θα αυξανόταν αν γινόταν μέλος και η Ελβετία. Ε, Όσον αφορά την, τις τρεις μικρές χώρες, αυτό θα, ε, η προσχώρησή τους θα διεύρυνε την ε, ευρωπαϊκή οικογένεια και θα βοηθούσε την ροή αγαθών ένα καλό παράδειγμα είναι η συνεργασία με την Ορβηγία. Πρόκειται για ε, ένα πρόγραμμα το οποίο διευκολύνει την ε, διαδικτυακή ε, διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών και κρατικών προμηθειών. Πιστεύω ότι ο χώρος αυτός εξάλλου θα έπρεπε να διευρυθεί και με την Τουρκία. Η Τουρκία είχε επί 50 χρόνια τώρα συμφωνίες σύνδεσης και ακόμα δεν έχει ε, άμεση, άσχεση, ε, άμεση πρόσβαση στην αγορά. Μια τέτοια πρόσβαση θα βοηθούσε την οικονομική ανάπτυξη και ίσως έχει έρθει η στιγμή ε, να ξαναδούμε την συμφωνία έχω ώστε να διορθώσουμε τα τυχόν κενά που υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επιτροπή, Χρόνια τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ασχοληθεί στην ολομέλειά του ζήτημα, με το ζήτημα της προσέγγισης των μικρών αυτών κρατών, Σαν Μαρίνο, Αγίου Μαρίνου, Ανδόρας και Μονακό. Και χαίρομαι που έχετε συμφωνήσει για τη συζήτηση του θέματος αυτού για χρόνια. Συζητούνται στους διαδρόμους ε, λύσεις για ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη αυτά είτε τα θέματα ήταν η φορολογία, είτε τα χρηματοπιστωτικά, βλέπουμε ότι έχουν κάνει σημαντικέ προσπάθειε τα κράτη αυτά για να μονοσυνήσουν την ε, νομοθεσία του με αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα τρία μαζί έχουν μόλις 150.000 κατοίκους. Τα μικροκράτη αυτά λοιπόν είναι συνήθως οι λησμονημένοι συγγενείς της εξωτερικής μας πολιτικής, που όμως έχουν ένα μαζί μας δεσμούς αρχαίους, ιστορικούς και καθημερινής συνεργασίας. Από τη Γαλλία εγώ γνωρίζω πολύ καλά το περικυπάτο της Ανδόρας, μια πολύ ισχυρή ε, παρουσία στη λειτουργία της ε, οροσυράς των Πυρηναίων και στην ιστορία της. Και όμως ε, υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά και δεν είναι εύκολο για τους κατοίκους της χώρας αυτής να εγκαθίστανται ή να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι επιχειρήσεις τους μπορούν να εισάγουν ή να εξάγουν τα προϊόντα τους. Το χειρότερο είναι ότι οι φοιτητές τους εκεί που μπορούν οι μη Ευρωπαίοι φοιτητέ να έρχονται με τα εράσμου, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αρθεί αυτό το εμπόδιο στην πραγματική ολοκλήρωση της ε, επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Έχουμε μία πρόταση για αξιολόγηση των προόδων ε, της Ανδόρας. Πρέπει να τηρηθούν βεβαίως οι προθεσμίες ώστε να μην αποθαρρυνθούν στις προσπάθειες τους οι μικροί μας αυτοί γείτονες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι είναι δυνατή η ολοκληρώση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και βέβαια καλό θα ήταν με μια πολύ προσεκτική, απλή, ανοιχτή, ειλικρινή και προς το συμφέρον όλων στην εργασία. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλστρομ για τις απαντήσεις της. Γιατί αποδεικνύουν ότι Πράγματι, η Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι χρήσιμη, χρειάζεται όμως να ε, διορθωθούν κάποια κενά ενδεχομένω. Η σχέση μας με αυτές τις χώρες πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και ταυτόχρονα στην αναλογικότητα. Δηλαδή, αφενός έχουμε από τη μια μεριά έχουμε μισό δισεκατομμύριο άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά έχουμε τρία μικροκράτη. Μιλούμε για διαφορετικές τάξεις μεγέθους. Χρειαζόμαστε όμως πρόσβαση στις αγορές αυτών των χωρών, έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να ε, δούμε όμως και ποια θα είναι η δική τους πρόσβαση στις δικές μας αγορές. Δεν θα σημαίνει βέβαια νουρίς αυτοκίνητο-βιομηχανίες οι χαλβουργικέ, αλλά σίγουρα είναι ισχυρά αυτά τα κράτη στην, στον τραπεζικό τομέα, παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα κράτη καταρχήν θέλουν να μπουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ε, Κυρίε και κύριοι, η εσωτερική αγορά προσφέρει ωφέλη στα κράτη-μέλη και τους πολίτες τους προσφέρει καταπληκτικές ευκαιρίες στην ελευθερία της κυκλοφορίας, στην ελευθερία της απασχόλησης σε μια άλλη χώρα, της εκπαίδευσης, οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει ε, και την, ε, στην εξέβρεση θέσης εργασίας, τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι δραστηριότητε λοιπόν μπορούν να απτυχθούν σε καλύτερους, σε περισσότερους ε, τομείς σε όλα τα κράτη-μέλη και να προωθήσουν έτσι τις θέσεις εργασίας. Έχουμε μεγάλες ευκαιρίες λοιπόν για οικονομική ανάπτυξη χάρη στην κινητικότητα και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των δεσμών με τις χώρες εκείνες όπως ο Άγιος Μαρίνος και το Μονακό που επιθυμούν να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευρύνουμε έτσι τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ε, προ όφελο όλων μα, γιατί διευρύνουμε το πεδίο των δραστηριοτήτων μα, τι ευκαιρίε για όλου μα. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για ε, συνεργασία με τα κράτη αυτά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι μία από τι επιλογέ, τι ευκαιρίε που έχουμε, τι εναλλακτικέ αν θέλετε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε πάνω απ' όλα του όρου τη συνεργασία και να ενισχύσουμε τις διατάξεις σχετικέ με την ενιαία αγορά. Ε, διαρωτώ με λοιπόν, ποια ε, στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει κατά προτεραιότητα να βελτιωθούν σε σχέση με τους κανόνες εσωτερικής αγοράς. Διότι αυτή τη στιγμή όταν εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ένα κράτος, οι διατάξεις σχετικέ με την εσωτερική αγορά γίνονται τμήμα της εσωτερικής του νομοθεσίας. Άρα πρέπει και η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής να καταστεί σημαντικό κομμάτι της συνεργασίας. Ο, κύριος, ο αντιπρόεδρος κύριος Κάρας έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς Επιτρέψτε να σας ευχηθώ και εγώ κυρία Πρόεδρε θερμά για τα γενέθλιά σας αυτή την εβδομάδα και δεύτερον να περάσω στο θέμα μας και το στόχο της συμφωνίας που ορίζεται και στο άρθρο πρώτο, που είναι μια πλήρης και ισορροπημένη ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συμβαλωμένων μερών, η ομοιογενής ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι μόνο των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, αλλά και στους λεγόμενους συμπληρωματικούς τομείς υπάρχει περιθώριο για συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και απαραίτητο διότι από καιρό έχουμε εντοπίσει ότι και στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη, τη γενική αλλά και την ειδική εκπαίδευση, την απασχόληση των νέων, την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα, είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι ένας με τον άλλον. Πρέπει λοιπόν, και το λέω ξεκάθαρα, να ξαναδιατυπώσουμε την έννοια Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, να αναλογιστούμε τι σημαίνει, τι συμπεριλαμβάνει και η Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά είναι η βασική ε, αρχή και προϋπόθεση της ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διπλανό εδώ κτίριο που βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και πρέπει να, να, να συζητούμε θέματα της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει ενταχθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης προηγουμένως και το ίδιο χωρίς να είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού, Χώρου, γιατί είναι ο προθάλαμος των διαδικασιών της ένταξης ε, το Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος στο οικονομικό πεδίο, όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πεδίο των δικαιωμάτων. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό όρο, Εάν τον εισαγάγουμε θα έχουμε κερδίσει πολύ χρόνο και κόπο και θα έχουμε ενισχύσει πολύ σημαντικά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Uh, Η κυρία τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από 21 χρόνια ε, υπογράφηκε η Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Χώρου που επέτρεψε η ενιαία αγορά να διευρυνθεί σε τρεις χώρες ΕΖΕΣ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Επέτρεψε επίσης οι οικονομικές και εμπορικές ε, σχέσεις ε, μεταξύ των δύο αυτών μερών να ενισχυθούν σε μια, μέσα σε μια ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της ενιαίας εσωτερική αγορά. Ε, όμως το 2012 η αξία των εμπορικών συναλλαγών ε, ήταν 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρόλο ότι η, ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει ε, συμπληρωθεί πλήρως. Σαν Μαρίνο Ανδόρα και Μονακό τώρα ζητούν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων και θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης που χρειάζεται τόσο πολύ η Ευρώπη. Περιμένουμε ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και στην επιπτώσεων που ε, γίνεται αυτή τη στιγμή και για την οποία μας μίλησε η Επίτροπος. Τελειώνω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιολογήσει, να αποφασίσει και να πράξει, να αξιολογήσει ε, τη λειτουργία ε, του οικονομικού χώρου και της συμφωνίας που το δημιουργήσε, να δράσει μειώντας τις αδυναμίες και τα κενά και δημιουργώντας προϋποθέσεις προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφασίσει για την ενίσχυση των σχέσεων με τις τρεις αυτές μικρές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προχωρούμε με το Catch the Eye. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον συνάδελφο Πλάνκοβιτ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ήθελα να... Ήθελα να πω ότι μια που έρχομαι από την ε, Κροατία, που μόλις προσχώρησε, ε, πρέπει να σας πω ότι και εμείς ε, ε, συμμετείχαμε στον ΕΟΧ και πρόκειται όσον αφορά τις χώρες ΕΖΕΣ για χώρες που είναι εντελώς ενταγμένες στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα η ένταξη του στον ΕΟΧ. Η Ισλανδία παρετήθηκε από το στόχο αυτό για διάφορους λόγους. Είμαι όμως ικανοποιημένο από την ανάλυση που έκανε η Επίτροπος Μάλστρομ σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία στα πλαίσια του ΕΟΧ και χαιρετίζω ιδιαίτερα τις ε, τρεις εναλλακτικέ λύσεις που ανέφερε η Επίτροπος για τις ε, χώρες αυτές που θα πρέπει να βρουν τη θέση τους στην συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και καθώς είμαι Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τι σχέσει με τον ΕΟΧ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω την Επιτροπή τη Ιστορική αγορά για την υποστήριξη στην προσπάθεια αυτή. Εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει η αναθεώρηση του ΕΟΧ να λάβει υπόψη τι εξελίξει στην εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, θέση σε εφαρμογή, την μεταφορά και την παρακολούθηση τη λειτουργία τη νομοθεσία τη εσωτερική αγορά. Είπε η, Ευρωπαϊκή, η ότι εδώ και 30 χρόνια έχουν αλλάξει τόσο πολλά. Η Ανδώρα, λοιπόν, ο Μαρίνο Μαρίνο στο Μονακό, είναι τρεις μικρές χώρες ε, με τις οποίες έχουν αναπτυχθεί ήδη συνομιλίες μέσω των ε, πρεσβευτών τους και συνεχίζονται. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος είναι κατάλληλο μέρος για την ανάπτυξη των ε, συνομιλιών. Βεβαίως περιμένουμε την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και για την Ελβετία, μια πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης πιστεύω μπορεί σε συνεργασία και με το Συμβούλιο αλλά και με το Κοινοβούλιο και πάνω στις κοινέ γραμμές που έχουμε ορίσει και με τις οποίες συμφωνούμε να ε, συμπεριλάβει έναν διακοινοβουλευτικό πυλώνα και να προβλέψει μια λύση η οποία θα επιτρέπει και στο Κοινοβούλιο να συμβαλάβει θελητικά. Ε, Ευχαριστώ και ο τελευταίος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Μάιλενβιτς. Η κυρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ΕΟΧ υπάρχει από το 1994 και έχει από τότε δώσει θετικά αποτελέσματα Παρόλε τις ε, αλλαγέ που μεσολάβησαν τα τελευταία χρόνια, διευρύθηκε η Ευρώπη και οι κανόνες ε, που ίσχυαν ε, στον ΕΟΧ άλλαζαν συνεχώς και φτάσαμε πάνω να έχουμε τώρα πάνω από 6.000 νόρμες, πρότυπα. Ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και για την ε, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα πρέπει να απαντήσουμε στα πλήγματα που δέχεται το σύστημά μας λόγω της κρίσης. Πρέπει να δείξουμε ελαστικότητα και να τροποποιήσουμε τους θεσμικούς μηχανισμούς και τα πρότυπα και να επιτρέψουμε μια πιο ορθολογική χρήση των εθνικών και ευρωπαϊκών προϋπολογισμών για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να μειώσουμε την ανεργία. Ευχαριστώ. Ε, Ήταν πολύ μακριά αυτή η μέρα. Ε, ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ορισμένε ερωτήσει για την Ελβετία. Για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει για την ενέργεια, ε, έχουμε διαπραγματεύσει για το θεσμικό πλαίσιο που θα πρέπει επίση να ολοκληρωθούν πριν ε, εφαρμοστεί οποιαδήποτε συμφωνία και οι συζητήσει αυτέ, οι διαπραγματεύσει αυτέ έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στην Ελβετία να συμμετάσχει στην εσωτερική αγορά με συγκεκριμένου όρου βέβαια σε ό,τι αφορά το θέμα του Σαν Μαρονίνο, την Ανδρά και το Μονακό, ε, εξετάζουμε διαφορετικά σενάρια, όπω είπα, στην έκθεση την οποία θα δημοσιεύσουμε σε δύο μήνε περίπου και θα τη συζητήσουμε μαζί σας. Ε, από νομική πλευρά για να είναι, γίνει κανεί μέλο του Ευρωπαϊκού Χώρου, θα πρέπει μπορεί να, αυτό να επιτευχθεί είτε μέσω συμμετοχή ε, ω μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσω της ΕΖΕΣ. και καμία αυτές τρει τρεις χώρες δεν έχει ζητήσει να γίνει μέλο τη ΕΖΕΣ, Οπότε ίσω θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση για να ικανοποιήσουμε αυτές τις τρεις χώρες. Και ο Μέσσερ Σμιτ, ναι. Ε, είναι ε, σημαντική πτυχή, η εξωτερική πτυχή της πολιτικής μας σε σχέση με αυτές τις τρεις μικρές χώρες. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση στις ανησυχίες σας. Τέλος για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Προφανώς είναι υποχρέωση οποιαδήποτε χώρα θέλει να συμμετάσχει στην ε, εσωτερική αγορά. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στην περίπτωση των τριών μικρών χωρών. Το αναλύουμε στην εκθέση που θα υποβάλουμε. Θα πάρετε λοιπόν περισσότερες απαντήσει. Ε, ενημερώστε την κυρία Στον για τις ανησυχίες σας αν θέλετε και θα επανέλθουμε και η κυρία Στον και εγώ σε δύο μήνες να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ για τη συζήτηση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι. Αύριο η επόμενη σύνο, περίοδο συνόδου στις 8.30 το πρωί. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ.